Σα Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Νταφ και σας ευχαριστώ όλους για αυτή την μακρά και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Η ψηφοφορία δεν θα γίνει σήμερα γιατί θα αναπαιμφθεί το θέμα στην Επιτροπή. Τώρα θα συζητήσουμε την έκθεση του κυρίου ε, Τζέφρεϊ Βαν Όρντεν για τη δράση κατά των ναρκών. Ο κύριος Βανόρντεν έχει το λόγο. Uh, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, λέει κύριος Βανόρντεν. Πρώτα πρώτα να σας πω ότι αισθάνομαι απογοήτευση γιατί δεν έχουμε τον χρόνο να συζητήσουμε πλήρως το σύμβολο αυτό θέμα ή στην Ολομέλεια ε, έχω συγκεντρώσει συνένεση ευρεία από όλες τις εταιρείες του Κοινοβουλίου και ευχαριστώ ε, για αυτό το λόγο όλους τους σκιώδες ηγητές. Όλα ξεκινήσαν δεκαετία του 90 ώστε να ε, μπει ένα τέρμα σε αυτές τις ε, νάρκες διότι χιλιάδες ζώων έχουν χαθεί από αυτές ε, κάθε χρόνο και επίσης έχουμε και άλλους οι οποίοι έχουν μείνει ανάπηροι για έχουν τραυματιστεί ε, αυτές οι ε, νάρκες κατά προσωπικού είπαμε πλέον να μην συγκαταλέγονται στους εξοπλισμούς του στρατού να γίνει μια τεράστια και έγινε κινητοποίηση πολιτική βούληση υπήρξε ε, πόροι στρατεύτηκαν από μη κυβερνητικού οργανισμούς γιατί μιλούμε για κάτι το οποίο όχι μόνο κοστίζει ζωές αλλά φρενάρει και την ανάπτυξη για κάποιες πάρα πολύ φτωχές χώρες που έχουν εμπλακεί σε ένοπλες αναμετρήσεις. Ε, ξεκινούμε επομένω να λαμβάνουμε υπόψη το πω αυτό το δύσκολο πρόβλημα θα επιληθεί. Όμως, γιατί δεν προχωρήσαμε πιο γρήγορα. Έχουν περάσει πάρα πολλά 14 χρόνια και έχουν πάνω από 90 χώρε οι οποίες ε, ακόμη ε, χρησιμοποιούν ή έχουν ως υπολείμματα τέτοιες ε, νάρκες κατά προσωπικού και ακόμη Έχουμε πάρα πολλού πόρου οι οποίοι δαπανώνται και αναλώνονται για αυτόν τον σκοπό. Επισύρουμε ακόμη μια φορά την προσοχή ει αυτό το πρόβλημα. Κατ' εξοχήν τα ευρωπαϊκά δεσμικά όργανα έχουν εμπλακεί σε αυτόν τον αγώνα. Θα πρέπει βεβαίω να χαιρετήσουμε του παθέ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί είναι πρωταγωνιστή σε αυτή την προσπάθεια. Αλλά και κάποια κράτη-μέλη. Η ΕΠΑ, ο Καναδά και άλλα κράτη βοηθούν πολύ. Οπότε, σε αυτή την ε, έκθεση για τις νάρκες λέμε για τις ε, ενάγκες κατά προσωπικού κυρίως, αλλά λέμε ότι ακόμα έχουμε και άλλες, ε, και άλλες νάρκες, νάρκες διασποράς κλπ. Οπότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι όλες οι δυτικές δημοκρατίες έχουν συστατευτεί. Προσπαθούμε, τα κίνητρά μας είναι καλόπιστα και δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι νιώθοντας ένοχοι θα βοηθήσουμε και Προσπαθούμε να αναδείξουμε κάποιες περιπτώσεις όπως η Μπούρμα, η Λιβύη, κάποιες ομάδες όπως ο ΦΑΡΚ. Αυτοί τις χρησιμοποιούν, άρχισαν να χρησιμοποιούν πρόσφατα ή φτιάχνουν τέτοιου είδους εκρητικούς μηχανισμούς. Πρόκειται για απειλή όχι μόνο κατά των ενόπλων δυνάμεων που αναμετρώνται, αλλά απειλείται και ο άμαχος πληθυσμός. Επομένως, ακριβώ προσπαθούμε να προστατεύσουμε αθώους πολίτες που πλήσονται στην καθημερινή του ζωή. Έχουμε σεμινάρια, έχουμε μια διεθνή εκστρατεία, έχουμε στη Γενέβη ένα ανθρωπιστικό μηχανισμό, έχουμε τον Ερυθρό Σταυρό που προσπαθεί, έχουμε ε, ένα διεθνές ίδρυμα που έχει έδρα την Σλοβενία για αυτές τις ε, νάρκες. Οπότε, και άλλοι έχουν βοηθήσει. Ε, έγινε αυτό το σεμινάριο και όλοι συμφώνησαν ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αφιερώσει ένα κονδύλι στην καταπολέμηση αυτών των ναρκών. Όμως, η οικονομική συγκυρία είναι δύσκολη. Οπότε, το μήνυμα της έκθεσής μου είναι ότι θα πρέπει να έχουν πιο στοχευμένη προσπάθεια, να βοηθήσουμε συγκεκριμένες χώρες περισσότερο και θα πρέπει να αποθαρρυνθούν χώρες που δεν τους περισσεύουν τα χρήματα να τα αναλώνουν για τέτοιες εκρηκτικές συσκευέ. Πολλές χώρες βέβαια στηρίζονται στη διεθνή βοήθεια. Θα μπορούσαν να βοηθήσουν περισσότερο. Υπάρχουν κάποια άλλα κράτη όπως η Βοσνία όπου σταμάτησε ο πόλεμος αλλά ακόμη έχουν απομείνει οι μηχανισμοί που εμποδίζουν την πρόοδο. Θα πρέπει επομένω να εκπαιδευτούν οι στρατιώτε στι χώρε για να γίνει απαραίτητη ναρκαλίευση. Εν κατακλείδη, σα επαναλαμβάνω πρόεδρε, ότι χρειάζεται περισσότερο συντονισμός, να κοιτάξουν ξανά τις προτεραιότητε μας, να υπάρξουν έρευνες, μελέτες για τη διαδικασία. Χρειάζεται πιο ευφυής κατανομή των πόρων για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο το οποίο μπορεί να καταπολεμηθεί. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια ρεαλιστική δυνατότητα που την έχουμε. Πρόεδρος, <clears throat> κύριε Φανόρντεν, σα ευχαριστούμε για την εισήγησή σα. και τώρα στα πλαίσια του Catch the Eye θα λέω το λόγο η κυρία Μπασέσκου. Θεωρώ ότι η έκθεση Van Orden ε, ασχολείται με ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ασφάλειας που πλήττει την Ευρώπη οι ε, μάρκες κατά προσωπικού χρησιμοποιήθηκαν ήδη από τους Βαλκανικούς πολέμους και βλέπουμε ότι το κόστος είναι μακροχρόνιο. Δεν διαθέτουν τα κατάλληλα κονδύλια όλα τα κράτη για να απομακρύνουν τις ε, νάρκες και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να ε, εκραγούν αυτές οι νάρκες. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει λοιπόν να γίνει η απομάκρυνση των ναρκών από τις πρώην εμπόλυμες ζώνες. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε και την συνδρομή των τοπικών αρχών. Θα ήθελα να κάνω έκκληση και στις εξειδικευμένες μη κυβερνητικέ για να ασχοληθούν με αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Η κυρία, η Κοπά έχει το λόγο. Ε, κυρία Πρόεδρε, οι σοσιαλιστές και δημοκράτες εκφράζουμε ικανοποίηση που 12 χρόνια μετά τη σύμβαση της Οτάβας μπορούμε να καταγράψουμε σημαντική μείωση των θυμάτων από νάρκες κατά προσωπικού. Και είμαστε περήφανοι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρωτοστάτησε και συνεχίζει να πρωτοστατεί στη διεθνή ε, προσπάθεια για έναν κόσμο χωρίς νάρκες όμως το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί και χιλιάδες άνθρωποι υποφέρουν ακόμα από τις συνέπειες αυτών των όπλων με την έκθεση που συζητάμε σήμερα προσπαθούμε να δούμε πώς θα βελτιώσουμε τη διεθνή μας δράση προκειμένου να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. είναι καιρός να ξαναδούμε τη συνολική εικόνα και να επιδιώξουμε μια δράση κατά των αρκών που να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερη συνεκτική και περισσότερο επικεντρωμένη στο συμφέρον των εμπλεκόμενων πληθυσμών. κατά συνέπεια η διεθνή και επιτόπου δραστηριοποίησή μα δεν πρέπει να καλύπτει μόνο τι νάρκες κατά προσωπικού αλλά και τα άλλα κατάλοιπα του πολέμου όπως τα πυρομαχικά διασποράς. ακόμα μεγαλύτερη έμφαση δε πρέπει να αποδίδεται στην εκπαίδευση και ενημέρωση των υποψηφίων θυμάτων που τις περισσότερες φορές είναι ανυποψία στα παιδιά. θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εισηγητή κύριο van orden για την εξαιρετική έκθεση που παρουσίασε αλλά και τη συνεργασία με όλους τους σκιώδεις εισηγητές καθ' όλη την εκπόνηση της έκθεσης αυτής. σας ευχαριστώ. Euh, Η κυρία έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα, σαν μια ψυχιώδη ηγετρίας, να ευχαριστήσω τον κύριο Φανόντον για την πολύ καλή αυτή συνεργασία και γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και εντάξατε πολλές ε, τροπολογίες, ε, πολύ καλή είναι η έκθεση τελικά. Λυπούμε που δεν έχουμε συζήτηση από αυτές. Θα ήθελα να θέσω το θέμα που παρουσιάστηκε μετά τη συζήτηση στην ΑΦΕΤ και γι' αυτό αυτό το θέμα δεν συμπεριλαμβάνεται. Τον Μάη μόλον, μία ένωση πολλών μη κυβερνικών οργανώσεων, Pax Christi κλπ. Δημοσίευσα μία έκθεση, θα σας τη δείξω εδώ, που αναφέρει το θέμα των επενδύσεων σε αυτού του τύπου τους οπλισμούς. Αναφέρεται στις ε, επιχειρήσεις, ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες και άλλες που χρηματοδοτούν την παραγωγή αυτών των ναρκών. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να σταματήσει, γιατί το επικρίνουμε και εμείς στην εκθεσία. Θα ήθελα να καλέσω όλα τα κράτη-μέλη, την Κομισιόν, το Συμβούλιο, όλα τα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία αυτών των μη κυβερνικών οργανώσεων, να μην υπάρχει πλέον οικονομική δέσμευση και χρηματοδότηση αυτών των όπλων. Ευχαριστώ κύριε Λούνα Τσέκλει. λέει η πρόεδρο. Ο κύριος Ομπερμάιερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκατό εκατομμύρια νάρκε κατά προσωπικού υπάρχουν ένα το κόσμο και κλασικά τα θύματα κατά 70% δυστυχώς είναι άμοχος πληθυσμό η σύμβαση της ΟΤΑΒΑ είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά και εμείς θα πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσουμε λίγο τα κράτη-μέλη γιατί το 66 χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπάρχουν παραδείγματος χάρη στην πόλη μου στην Λίντς 700 βόμβες αεροπορικές που δεν έχουν ακόμα εκραγεί και το κόστος που είναι πάρα πολύ υψηλό για την εξάρτησή τους το φέρουν οι ιδιοκτήτες των κτηρίων στο οποίο βρίσκονται οι βόβες αυτές. Γι' αυτό στρέφουμε προς την Ευρωπαϊκή Κομισιόν. Γιατί εδώ νομίζω δεν κάνουμε αυτό που ε, πρέπει. Θα πρέπει να, ε, ε, να γνωρίζει το πρόβλημα αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν το γνωρίζει φαίνεται. Ευχαριστώ κύριο Σκέλαμ. Thank you very much, Ευχαριστώ ο συνάδελφος ε, Βαν Όρντεν μας ε, έδωσε μία επίκαιρη ε, έκθεση μετά από ένα σεμινάριο που έγινε επί του θέματος. Η έκθεση δακτυλοδεικτεί ορισμένες χώρες οι οποίες ε, απομακρύνθηκαν από τον κατάλογο χριστών μόλις πέρσι. Και γίνεται λόγος και για την Κίνα και τη Ρωσία που έχουν μεγάλα αποθέματα. 124 εκατομμύρια δηλαδή νάρκες κατά προσωπικού. Η έκθεση καταδεικνύει ότι ορισμένες χώρες βασίζονται στη διεθνή βοήθεια. Θα πρέπει οι ίδιες οι χώρες να αναλάβουν ε, την ευθύνη και να εκαθαρίσουν τις ε, περιοχές τους από τις νάρκες. Επίσης θα πρέπει να βοηθήσουμε τα θύματα. Πρόκειται για ένα μακροχρόνιο αγώνα και θα πρέπει να υπάρξει ε, διεθνής αλληλεγγύη βεβαίως με τη χρηματοδότηση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έληξε ο γύρος Catch the και δίνω το λόγο στην ε, κυρία Επίτροπο για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Ευχαριστώ. Αγαπητά μέλη του Συμβουλίου, καλωσορίζουμε την πρόοδο με βάση την έκθεση του κυρίου Βαν Όρτεν για τις νάρκες κατά προσωπικού. Θεωρούμε ότι έχει επιτελεστεί πρόοδος. παρόλα αυτά, πολλά πρέπει να γίνουν ιδιαίτερα σε σχέση με τις πλέον ευάλωτες χώρες, οι οποίες χρήζουν διεθνούς βοήθειες και να βοηθήσουμε και τα θύματα βεβαίως θα πρέπει να εξαλειφθούν οι νάρκες κατά προσωπικού και να αναφερθούμε και στα συναφή οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Η έκθεση τονίζει ότι αν και τα νέα θύματα μειώνονται, ο αριθμός τους μειώνεται, παρόλα αυτά χρειάζονται αρρωγή τα θύματα αυτά. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις προκλήσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Η έκθεση ασχολείται με την μεγάλη προσπάθεια που έχει καταβληθεί από τη διεθνή κοινότητα. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη συλλογικά συνέδραμαν και με χρήματα και με την έρευνα για την απομάκρυση των ναρκών κατά προσωπικού. Η χρηματοδότηση έφτασε στο 1,8 δις ευρώ τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτό αποτελεί το ίμιση της διεθνούς χρηματοδότησης για την καταπολέμηση των και εξάλληψη των ναρκών. Μέσα στα πλαίσια των ε, κοινών δράσεων της εξωτερικής πολιτικής έχουμε ε, υποστηρίξει την εκαθάριση από τις νάρκες με βάση τη σύμβαση της ΟΤΑΒΑ και προωθήσαμε την ασφάλεια έτσι ώστε να προσχωρήσουν ακόμα περισσότεροι στη σύμβαση. Επίσης προετοιμάζουμε μία νέα απόφαση του Συμβουλίου μετά από την ε, δεύτερη αναθεώρηση της σύμβασης της ΟΤΑΒΑ μετά την ε, διάσκεψη της Καρταχένα στην ε, Κολομβία το 2009. Συνεισφέραμε κατά 400 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2002-2010. Τρίτον, συμφωνούμε ότι είναι αναγκαίο να αναθεωρήσουμε τις κατευθυντηρίες γραμμές για την κοινοτική δράση, έτσι ώστε να υπάρξουν εθνικά προγράμματα ανάπτυξης και ε, η διασύνδεση θεμάτων ασφαλείας και αυτού του προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι ότι οι χώρες που θα ευεργετηθούν θα θέσουν ως πρωταρχικό στόχο την εκαθάριση από τις νάρκες. Επίσης θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη αρρωγή και εθνική ανταπόκριση τουλάχιστον για τις χώρες που δεν μπορούν από μόνες τους να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Θα ήθελα να πω σε όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου ότι μέσω του μέσου σταθερότητας έχει γίνει μερική χρηματοδότηση και προβάλαμε και ανθρωπιστική βοήθεια στο βόρειο νότιο ε, Σουδάν, Πακιστάν και Σρι Λάνκα. Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω μία βασική πτυχή του θέματος που δεν καλύπτεται από την έκθεση. Μας απασχολεί όλο ένα αυξανόμενος αριθμός θυμάτων από νάρκες που έχουν εγκατασταθεί από μη κρατικούς ή εθνικούς φορείς. Θεωρούμε ότι θα πρέπει όλα αυτά να ενταχθούν στη σύμβαση της ΟΤΑΒΑΣ και θα ήθελα να σας τονίσω ότι αυτό, αυτή η πολιτική μας θα αποτελέσει προεξάρχον στοιχείο της πολιτικής της ΕΕ. Ευχαριστούμε την Επίτροπο. Λίγη, μάλλον διακόπτεται η Σύνοδος μέχρι τις 12 που θα γίνουν οι ψηφοφορίες.